προσαρμοστούμε στις δημογραφικές αλλαγές και θα προσδιορίσουμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία ε, ανάμεσα στα τρία αυτά τα μία. Ευχαριστούμε. Τελειώσαμε την έκθεση West, ε, West Lab και τώρα ξεκινάμε το τελευταίο σημείο. Την έκθεση Simon, κρατικές ενισχύσεις της Υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος. Ο εισηγητής παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ο βασικός πυλώνας του ευρωπαϊκού, του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και δεν παίζουν μόνο καθοριστικό ρόλο για τον μεμονωμένο πολίτη, αλλά έχουν μια τεράστια σημασία για την ευημερία του, του συνόλου της κοινωνίας, κατά την επεξεργασία της ε, ε, οδηγίες για τις κρατικές ενισχύσεις ε, για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος θα πρέπει να βρίσκεται στο προσκήνιο το εξή ερώτημα. Πώς θα πρέπει να διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για να έχουμε από τη μία μια υψηλή ποιότητα αυτών των υπηρεσιών και από την άλλη μια καθολική πρόσβαση για όλα τα τμήματα του πληθυσμού. βασικό στοιχείο για την οργάνωση ποιοτικά υψηλών υπηρεσιών είναι από τη μία η ασφάλεια των παρόχων και των δημόσιων αρχών όσον αφορά τις νομικές προϋποθέσεις πλαίσιο και από την άλλη μια ισχυρή αναλογικότητα των κανόνων, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές των διαφόρων ε, τύπων ε, υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και με τον τρόπο αυτό να μειώνεται το διοικητικό άχθος. Η μεταρρύθμιση των διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις μπορεί να γίνει λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη λειτουργία των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και τηρώντας αυστηρά την αρχή της επικουρικότητας. Για ένα επαρκές μέτρο νομικής ασφάλειας θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες υπηρεσίες. Νομική βάση θα ήταν για μας ε, τους Σοσιαλδημοκράτες το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ωστόσο εδώ δίστανται οι απόψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως γνωστόν εδώ και πολλά χρόνια και υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις. Παρ' όλα αυτά ε, πετύχαμε εμείς να εκπονήσουμε έναν συμβιβασμό ικανοποιητικό για όλες τις πλευρές. Οι αντισταθμιτικές πληρωμές για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα υψηλές. Αυτό ισχύει περισσότερο για μικρούς παρόχους υπηρεσιών η αύξηση των τιμών κατοφλίων για την απελευθέρωση από την υποχρέωση κοινοποίηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνοντας, ε, στην περίπτωση των κρατικών ενισχύσεων θα αποτελέσει μια πρώτη διευκόλυνση. Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να δημορφωθούν κατά τρόπο που το διοικητικό άχθος των τοπικών αρχών και των παρόχων ε, υπηρεσιών να βρίσκονται σε μια κατάλληλη αναλογία με τις ενδυνάμει επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή εξωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό. Οι προταθήσεις ε, ειδικέ de ε, ρυθμίσεις, δηλαδή μια γενική εξαίρεση από τις διατάξεις για τους τοπικούς παρόχους καθώς και για τις κοινωνικές υπηρεσίες αποτελούν μια σημαντική βάση για να δικαιώσουμε το ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών ζητούμε τον επαρκή ορισμό του χαρακτήρα τους και την προστασία τους. Επιπλέον με την έκθεση αυτή υποβάλλουμε την ε, πρόταση ή μάλλον εξτάζουμε την πρόταση τη Επιτροπής να υπάρξουν κριτήρια αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη συμβατότητα με τους ε, ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού. Αλλά εμεί το απορρίπτουμε αυτή την πρόταση τη Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι επιφερτισμένη μόνο με τον έλεγχο των ε, κρατικών ενισχύσεων. Η εφαρμογή των κανόνων εναπόκειται στις χώρες ε, μέλη και μπορεί να ρυθμιστεί μόνο με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό να κλείσω και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στην Επιτροπή, ιδιαιτέρως τους και ηγητές. Η ξεκάθαρη υπερψήφιση της έκθεσης στην Επιτροπή ε, αποδεικνύει αυτή την εξαιρετική συνεργασία που είναι προσανατολισμένη στην επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος. Είμαι σίγουρος αύριο στην ψηφορία στην Ολομέλεια θα πετύχουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για βιώσιμες προποθέσεις πλαίσιο στο τομέα των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ε, συμφέροντος. Ευχαριστούμε πολύ, ε, Σίμων. Και τώρα ε, θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Μεσάρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για τις ε, υπηρεσίες ε, γενικού συμφέροντος ε, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να είναι ανεξαρτήτως οδήματος προσβάσιμες για όλους τους πολίτες. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από οργανισμούς οι οποίοι δέχονται κρατικές επιδοτήσεις. Φυσικά πρέπει να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Φυσικά οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη εξισιοδότηση ώστε να οργανώνουμε σωστό τρόπο ε, την παροχή υπηρεσιών οι οποίες είναι και πάρα πολύ σημαντικές για την τοπική οικονομία και δημιουργούν πολυάριθμες θέσεις απασχόλησης. Χρειάζεται βελτίωση της υποδομής Όλο ιδιαίτερο δε στι περιοχές όπου παρατηρούνται οι βασικότερες ατέλειες. Χρειαζόμαστε ποιοτικέ υπηρεσίες, αποτελεσματική χρήση των πόρων σε προσιτέ για όλους τους καταναλωτές τιμέ. Αφετέρου χρειαζόμαστε καλής ποιότητας χώρους εργασίας. Ευχαριστούμε κύριος ε, Ντεκάμπος. Ευχαριστώ πρόεδρε, επίτροπε. Αυτή η έκθεση του συναδέλφου Πίτερ Σάιμον ε, είναι ιδιαίτερα ισοσκελισμένη. Χρησιμοποιεί τις ε, υπηρεσίες ε, γενικού συμφέροντος, όχι μόνο προβάλλοντας τις ως βασικές αξίες, αλλά και ως κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Υπάρχει φυσικά μία νομοθετική υποδομή, αλλά χρειαζόμαστε και ασφάλεια δικαίου και τήρηση της αρχής επικουρικότητας. Θετικά στοιχεία έχει η έκθεση η διάκριση ανάμεσα στι οικονομικέ και μη δραστηριότητε, η αναφορά ε, στα τοπικά και περιφερειακά επίπεδα που δεν επηρεάζονται την αγωνιστικότητα στην εσωτερική αγορά, η αναφορά ε, στα ομόλογα έργα, η αναφορά στου κανόνε εντεμήνυμη ε, και περιορισμό των κρατικών επιδοτήσεων. Τώρα, σε σχέση με το καταστατικό των παρόχων, καλύπτονται οργανώσει, σωματεία, μη κυβερνητικέ οργανώσει ενώσεις, είναι αρκετά εύρης ορισμός. Επίσης, ε, το θέμα της ασφάλειας του δίκαιου θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθεί με την τήρηση της αρχής επικουρικότητας. Αυτά και ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, ο κύριος Πάσκουα. Πρόεδρε, μέχρι το τέλος του 2011 πολλά μέτρα θα, πάβουν, να, θα πάψουν να ισχύουν. Μέτρα που αφορούν τις κρατικές ενισχύες. Επομένως είναι απαραίτητο να, να μεταρρυθμίσουμε αυτούς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Ε, με τους τρέχοντες κανόνες ε, πάρα πολύ οι τοπικές αρχές, ε, ε, υπήρχε τρομερό γραφειοκρατικό άχθος και επίσης δεν υπήρχε ασφάλεια δικαίου. Η μεταρρύθμιση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων θα φέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι κανόνες θα πρέπει να είναι πιο απλοί, πιο εύκολοι στην εφαρμογή τους ούτω ώστε και σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο να μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά. Αυτό νομίζω θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ε, υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, αξιότιμε κύριε Πίτροπε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πέτερ Σίμων για το πώς πραγματικά εργάστηκε ξεπερνώντας τα όρια μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Και ε, κατόρθωσε να καλέσει την Επιτροπή μέχρι το 2012 να υποβάλει μία δήλωση συμπεριλαμβάνοντας κάποια μέτρα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο είπε ήδη ο κ. Σίμαν. Φυσικά θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά το 2014 να συμβάλλει στην νομοθετική διαδικασία. Η Επιτροπή ζητά από όλους ενεχόμενους διαφάνεια, διαφάνεια, διαφάνεια και ε, αντίθετα στην πράξη προσπαθεί ε, με επισπεσμένες διαδικασίες μέσω της ε, διαμόρφωσης, ε, να περάσει τις δικές της απόψεις. Η Ευρώπη ζει στο επίπεδο των περιφερειών και είναι εντυπωσιακό ότι ειδικά οι άνθρωποι στις περιφέρειες και στους τοπικούς φορείς γίνονται πολύ συχνά αντικείμενα επίθεση από την Κομισιόν ή περιθωριοποιούνται με αυτό το πλαίσιο ε, θίγεται το θέμα αυτό ε, και θα ήθελα να υπενθυμίσω τη βασική αρχή ενωμένη στην ε, πολυμορφία United and Diversity ε, καλώντας την Επιτροπή να στηριχθεί στο άρθρο 14 και τη δυνατότητα συνύπαρξης η κυρία Ρόιτοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στον τρόπο που προσδιορίζουν την εμβέλεια των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και τις εξαιρέσεις από τους κανόνες. Πρέπει να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προσπάθειες ε, να χαρτογραφήσει τις, ε, τις μεθόδους των κρατών μελών. Θα πρέπει να πλουστευτούν οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων και να υποστήριξουμε την Κομισιόν στην προσπάθειά της να εισαγάγει μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο με σεβόμενη βέβαια την αρχή των, της επικουρικότητας. Ε, οι μεγάλες επενδύσεις σε, για τοπικές συμβάσεις ενέχουν τον κίνδυνο μεγάλης διαφθοράς. Υπάρχουν πολλές, πολλά προβλήματα διαφθοράς εκεί. Επίσης θα πρέπει η Κομισιόν να μπορεί να ε, ελέγχει ε, οποιασδήποτε υπόνοιες για προβλήματα. συχνά γίνονται επίσημοι έλεγχοι επίσημες, επίσημες έρευνες χρησιμοποιώντας ε, τις πληροφορίες που δίνουν ε, αξιωματούχοι της κυβέρνησης οι οποίοι αποπειρώνται συχνά να κρύψουν ε, παρατυπίες σε σχέση με τους κανόνες των κρατικών ισχύσεων. Ευχαριστώ. Οι υπηρεσίε γενικού οικονομικού συμφέροντο ε, αυξάνουν την ευημερία και την οικονομική ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών. Αυτέ οι υπηρεσίε είναι σημαντικέ για την καταπολέμηση των ε, κοινωνικών ανισοτήτων. Η αντιστάθμιση για αυτέ τι ε, υπηρεσίε δεν πρέπει όμω να διασαλεύει τον ανταγωνισμό και δεν θα πρέπει να πλήττει άλλε επιχειρήσει. Θα πρέπει να γίνει σεβαστή η αρχή τη επικουρικότητα ε, το πρωτόκολλο 26 της ε, Συνθήκης της Λισαβόνας. Βάσει αυτού, τα κράτη-μέλη έχουν ε, αρμοδιότητες για να εξασφαλίσουν τις δημόσιες υπηρεσίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Στη Ρουμανία αυτοί οι κανόνες θα πλουστευτούν για τις δημόσιες υπηρεσίες σε περιορισμένη κλίμακα σε τοπικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστήξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να εξυγχρονίσουν τις ε, υπηρεσίες αυτές γενικού οικονομικού συμφέροντος και να τις προσαρμόσουν στις ανάγκες του κοινού. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένη νομοθεσία για κάθε τομέα στα κράτη-μέλη, κάθε τομέα αυτών των υπηρεσιών. Ε, κάποιος άλλος, νομίζω ότι σας βλέπω όλους. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε εκ μέρου του Αντιπρόεδρου κυρίου Αλμούνια. Ευχαριστώ τον κύριο Σάιμον για την έκθεσή του για τη μεταρρύθμιση των κανόνων κρατικών ισχύσεων για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Ε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εικόν και Ήτρε, καθώς και τα μέλη τους για τις συνεισφορές τους σε αυτή την έκθεση. Είμαστε επιπλησμένοι ότι οι δημόσιες υπηρεσίες είναι σημαντικές για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, γιατί συνεισφέρουν σημαντικά στην κοινωνική σταθερότητα και στην εδαφική συνοχή. Ακριβώς γι' αυτό οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων ε, και είμαστε ικανοποιημένοι που γίνεται τόσο έντονη συζήτηση για αυτό το θέμα μεταξύ των ε, Ευρωβουλευτών, άλλων θεσμικών οργάνων και των ενδιαφερομένων. Καλωσορίζουμε τη συνεισφορά του Ευρωκοινοβουλίου σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δείχνει τη σημασία που δίνει το Κοινοβούλιο στη δημιουργία ε, ενό αφού νομικού πλαισίου για τι ε, υπηρεσίε γενικού οικονομικού συμφέροντο. Να συμπενθυμίσω ότι η μεταρρύθμισή μα βασίζεται σε τρει στόχου. διευκρίνηση, απλούστευση και μια πιο πολυσχεδή προσέγγιση. Στην ανακοίνωσή μας του Μαρτίου ε, παρουσιάσαμε αυτού του στόχου αναλυτικά. Επίσης, ε, έκτοτε ετοιμάσαμε ένα κείμενο για να εξηγήσουμε πώς εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι αρχές. Ε, αυτό το κείμενο ήταν πλούσιο. Η κατεύθυνση της μεταρρύθμισης βρίσκει σύμφωνο σχεδόν όλους. Όλοι βέβαια οι φορείς έχουν διαφορετικές απόψεις για τις λεπτομέρειες των αλλαγών. Γι' αυτό ακριβώς σε επόμενε εβδομάδε θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε περισσότερο το πώ θα εφαρμοστούν, τον τρόπο εφαρμογή αυτών των στόχων. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήρθε πραγματικά ε, την κατάλληλη στιγμή. Γιατί έλαβε υπόψη το σχέδιο κειμένου μα και επομένω να κάνει και προτάσει για το πώ θα βελτιώσουμε περαιτέρω τα κείμενά μα. Ε, νομίζω ότι θα είναι πολύτιμο εργαλείο ε, για τη μεταρρύθμιση. Θα ήθελα σύντομα να εστιάσω σε τρία ε, σημεία της έκθεσης Σάιμον. Ένα βασικό εργαλείο για την απλούστευση στη μεταρρύθμισή μας είναι το, ο νέο κανονισμό de minimis, ελαχίστων προτύπων. Η έκθεση λέει ότι ένα κατόφλι που θα βασίζεται στο μέγεθος της κοινότητας δεν είναι απαραίτητο για να περιοριστεί ο κανονισμό de minimis ε, και μια ε, τριετής προσέγγιση είναι καλύτερη από την, ε, από την ισχύουσα μονοετή. Ε, θέλουμε να δούμε τι κατόφλια είναι πιο κατάλληλα. Ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει. Θέλουμε να μα πείτε ποιε είναι οι απόψει σας, ποιε είναι οι απόψει όλων των ενδιαφερομένων φορέων και κυρίω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βεβαίω. Δεύτερον, η έκθεση ζητάει ε, επιπρόσθετε κοινωνικέ υπηρεσίε να καλυφθούν από την απόφαση. Οι υπηρεσίε ε, κοινωνικού, ενδιαφε... Ε, παίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία μα. και πρέπει οπωσδήποτε να τι ελέγξουμε εκ του σύνεκης. Γι' αυτό ε, υπό την πιο πολυσχεδή αυτή προσέγγιση ε, εποφελούνται από την εξαίρεση ε, από την κοινοποίηση και πιο χαλαρά κριτήρια από αυτά που προβλέπει η απόφαση. Θέλω να αξιολογήσω οποιοδήποτε επιχείρημα για να βελτιώσω την ε, μεταχείριση των κοινωνικών υπηρεσιών, όπου αυτό βέβαια είναι απαραίτητο. Τρίτον, το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η Κομισιόν μπορεί να προωθήσει κάποια κριτήρια αποτελεσματικότητα στους κανόνες ε, κρατικών ενισχύσεων. Η Κομισιόν δεν τσεκάρει αυτή τη στιγμή την αποτελεσματικότητα. Το κείμενο, το σχέδιο κειμένου λέει ότι οι επιχειρήσει θα έχουν ε, κίνητρα για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά του. Ξέρω ότι ορισμένοι από εσά φοβούνται ε, τι ε, επερχόμενε αλλαγέ. Όμω τα κίνητρα αποτελεσματικότητα ισχύουν μόνο σε μεγάλου εμπορικού φορεί που αξιολογούμε μέσα στο πλαίσιο. Ε, Επίση, υπάρχει υπηρεσιών, υποστηρίζουν αυτά τα κριτήρια και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Θέλω να υπενθυμίσω ξανά ότι θέλουμε να βελτιώσουμε του κάμνες μα. Γιατί? Γιατί σήμερα που έχουμε τόσου περιορισμού δημοσιονομικού ε, και σε όλα τα κρατη που υπάρχουν τόσα προβλήματα, θέλουμε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να απολάβουν ε, ε, προσιτών και αποτελεσματικών ε, δημοσίων υπηρεσιών. Ακριβώ γι' αυτό. Αυτά και σα ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την πολύτιμη συνεισφορά σα στην έκθεση. Και εμεί σα ευχαριστούμε, Επίτροπε Νταλή, για την συνεισφορά σα και την παρουσία σας ε, εδώ στο Κοινοβούλιο σήμερα. Θα ψηφίσουμε αυτή την έκθεση του Πίτερ Σίμον ε, αύριο στι 12. Κλείνει η σημερινή συνεδρίαση. Θα τα ξαναπούμε αύριο.